Καλησπέρα. Θα αρχίσουμε, κυρίσω την άναρξη της συνεδρίασής μας. Είμαι προσωρινή πρόεδρος, προκειμένου να εκλέξουμε τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζω και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη σε αυτήν την συνεδρίαση συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής μας. Όπως γνωρίζετε, στόχος είναι να δημιουργήσουμε το Προεδρείο της Επιτροπής μας, να κλέψουμε δηλαδή τον Πρόεδρο και τους τεσσάρες αντιπροέδρους σύμφωνα με το άρθρο 204 του κανονισμού. Η σειρά είναι εξή. Πρώτον, Πρόεδρος και εφόσον έχει εκλεγεί ο Πρόεδρος, στη συνέχεια ο Πρόεδρος ή η Πρόεδρος θα αναλάβει την Προεδρία και θα ακολουθήσει η εκλογή των αντιπροέδρων. Ποιοι είναι αναπληρωματικοί που συμμετέχουν στην ψηφοφορία σήμερα, θα σας πω τώρα. ποιοι μα είπαν ότι αντικαθιστούν τακτικά μέλη. Μαρινέσκου από το ΕΛΚ για τον κύριο Πρεντά. Κονσάλ Λεγκρίπ, Κωνσταντς Λεγκρίπ, παρικαθιστά Βέκελ. Μπροκ, τον Μαλινόφ και η κυρία Κρέσλ, τον κύριο Σύριο. Σοσιαλιστές. Μανίκη, αντικαθιστά τον Ροζιέ. Από το Ευθέρη, κυρία Τινάσκα, αντικαθιστά την κυρία Θοχάρους, εκ μέρους του ΕΦΔΕ η Λάουρα Αγγία, αντικαθιστά τον Νταβίτ Κόμπουλ. Καλώς. Υπάρχει απαρτία. Σωστά. Για να δούμε. Για να είναι έγκυρη ψηφοφορία πρέπει να ψηφίσει το 1 τέταρτο των μελών της Επιτροπής μας. Η γραμματεία ελέγχει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τα τακτικά μέλη, αναπληρωματικά, απαρτία, ότι υποψήφοι έχουν υποβάλει την δήλωση οικονομικών του συμφερόντων επίσης. Ωραία, τώρα. Ποιοι είναι υποψήφοι για την θέση του Προέδρου της Επιτροπής μας. Παρακαλώ. Ελεονόρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους. Από πλευράς EFDD θα ήθελα να σας παρουσιάσω την υποψηφιότητα της Ελεονόρα Εύη, της ε, συναδέλφου, υποψηφιότητα για την Προεδρία της ε, Επιτροπής μας, σύμφωνα με τη μέθοδο DONT. Και σας ευχαριστώ. Άλλοι υποψήφοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Άλντε, θέλω να προτείνω την κυρία Σεσίλια Βίλκστρομ στη θέση της Πρόεδρου. Μαργαρέτα, ένα διαδικαστικό. Θέλω να πω σε όλους τους παρευρισκομένους ότι αν αγνοήσουμε πάλι το σύστημα DONT, τότε διακυδεύεται η δικαιοσύνη και η ειλικρίνεια στο σώμα καταλαβαίνω ότι μπορεί να χάσουμε, αλλά για την αξιοπρέπεια της ε, αντιπροσωπευτικότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το να μην δεχόμαστε το σύστημα αντών, το όπως έγινε πριν από δύο χρόνια, δεν είναι καλό. Ας καθίσουμε και ας σκεφτούμε αν αυτό γίνει συνήθεια και τελικά οι δύο μεγάλες ε, ομάδες μεταξύ τους ε, τα βρίσκουν και αποκλίνουν όλους τους υπόλοιπους. Αυτό ήθελα να υπενθυμίσω, τίποτα άλλο. Bien, Πρόεδρος, καλώς. Συνεχίζουμε με τη διαδικασία. Έχουμε δύο υποψηφιότητες. Μυστική θα είναι η ψηφοφορία. Έχουμε δύο υποψήφιες λοιπόν. Και σύμφωνα με τους κανόνες, μία ψήφο έχει ο κάθε βουλευτής. Και σύμφωνα με την κατανομή, η ΕΛΚ 10, σοσιαλιστές 8 ψήφους, 4 τη ΣΥΑΡ, 3 η ΑΛΔΕ, 3 ε, η ΓΚΟΕ, 2 ψήφους και το ΕΝΗ μία ψήφο. Στον πρώτο γύρο, όποιος υποψήφιος έχει την απόλυτη πλειοψηφία, κηρύσσεται νικητής. Αλλιώς υπάρχει δεύτερος γύρος. Εκεί περνάει όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας ο περισσότερο ηλικιωμένος υποψήφιος κερδίζει. Μυστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά θα γίνει. Έχετε την ηλεκτρονική σας κάρτα, φαντάζομαι, όλοι όσοι πρόκειται να ψηφίσετε σωστά. Καλώς. Θα σας εξηγήσω τώρα λίγο Πώ θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Υπάρχουν λοιπόν δύο υποψήφοι, είπαμε, η Σεσίλια Βίλστρομ και η Ελεονόρα Εύη. Θα δώσω ένα χρώμα στην κάθε υποψήφια και θα ψηφίσουμε ε, βάσει των χρωμάτων αυτών. Το πράσινο κουμπί είναι για τη Σεσίλια Βίλστρομ και το κόκκινο κουμπί θα είναι για την Ελεονόρα. Το άσπρο είναι για την αποχή, για όποιον δεν θέλει να ψηφίσει. Οπότε, ψηφίζουμε. Επαναλαμβάνω. Πράσινο κουμπί για την Σεσίλια Βίλστρομ και κόκκινο κουμπί για την Ελεονόρα Εύη. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Το ΕΛΚΑ έχει έναν παραπάνω που ψηφίζει από όσους επιτρέπεται. Εντάξει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Είκοσι ψήφοι υπέρ της Εσίλιας Βίλστρομ και 7 ψήφοι υπέρ της Ηλονόρας Εύη. Συγχαρητήρια. Δεν χρειάζεται δεύτερος γύρος, οπότε πρόεδρος μας είναι η Σεσίλια που θα έρθει εδώ στο Δήμο και θα αναλάβει την Προεδρία. Συγχαρητήρια πάντως και στις δύο. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Για μένα είναι πραγματικά τιμή που επανεξελέγει στην Προεδρία της Επιτροπής αυτής. Να ξέρετε ότι θα συνεχίσω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να λαμβάνω υπόψη όλους σας, όλες τις πολιτικές ομάδες και να είμαι πραγματικά πρόεδρος ολόκληρης της Επιτροπής αυτής, εκ μέρους των πολιτών της Ευρώπης των πολιτών που φτάνουν σε εμά με τα προβλήματά τους, με τα παράπονά τους, με τις ανησυχίες τους. Οπότε σας ευχαριστώ και πάλι και θα συνεχίσω το έργο μου να κάνω ό,τι μπορώ, να μην προεδρεύω τόσο, περισσότερο να σας εξυπηρετώ εσάς τους συναδέρφους. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ψηφοφορία και ερχόμαστε στην Αντιπροεδρία των Αντιπροέδρων. Ελεονόρα Εύη, ζητήσατε το λόγο. Παρακαλώ. Σεσίλια, σε ευχαριστώ. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να υποβάλω μια μικρή παρατήρηση όσον αφορά την ψηφοφορία, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ στενάχωρο το ότι για δεύτερη διαδοχή φορά μέσα σε δυόμιση χρόνια είναι κάτι το οποίο επαναλήφθηκε, κάτι το θλιβερό, κάτι το στενάχωρο. Δεν ξέρω εάν ετηρήθη τελικά η μέθοδος don't. Το σύστημα το οποίο όπως είπε η κυρία Όκεν είναι αναγκαίο ούτως ώστε να υπάρχει δίκαιη και αναλογική αντιπροσώπευση όλων των πολιτικών ομάδων, ιδίω δε των μικρότερων. Ισότητα είναι η λέξη κλειδί. Αυτή η υπέροχη λέξη που όμως τώρα δεν ίσχυσε. Τι να σας πω, αυτά τα δυόμιση χρόνια αποτελούν προηγούμενο για το κοινοβουλευτικό μας έργο, για μας σαν πολιτική ομάδα, σαν ε, ε, κόμμα των πέντε αστέρων, κίνημα των πέντε αστέρων. Σπάθατε με, αλλά σήμερα, συνάδελφοι, και οι άλλοι του FDD και το προσωπικό μας, με μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και να κατοχυρώσουμε ό,τι κατακτήσεις έχουμε κάνει σε αυτό το επίπεδο. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται όσον αφορά την κατανομή των θέσεων. Θα πρέπει να γίνει με αυτό το σύστημα το οποίο όμως παρεβιάστη, δεν ε, ίσχυσε. Γι' αυτό σας είπα για την ισότητα. Είναι υπέροχη λέξη για την πολιτική και γενικότερα. Οπότε η Επιτροπή των Αναφορών είναι η Επιτροπή που πρέπει να αφουγκράζεται όλους τους πολίτες και αυτό να γίνεται με την αρχή της ισότητας. Τέλος πάντων, όλες μου οι ευχές, συνάδελφοι σε όλους και στην Πρόεδρο. Και εγώ θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου, όπως πάντα, στην Επιτροπή μας. Thank you, Ευχαριστούμε, Ελεονόρα. Ας ε, το συζητήσουμε αυτό κάποια άλλη στιγμή, μια που τώρα είμαστε μέσω ψηφοφορίας. Είναι μια συνεδρίαση συγκρότηση σε σώμα, οπότε πρέπει να εκλέξουμε τους αντιπρόεδρους τώρα της Επιτροπής. Οι αναπληρωτές παραμένουν οι ίδιοι, έτσι, όπως και στην προηγούμενη ψηφοφορία. Η απαρτία επίσης την έχουμε. Οπότε, υποψηφιότητες για την πρώτη αντιπροεδρία. I Οι λοιπόν, για την πρώτη αντιπροεδρία, παρακαλώ. Ο Πίτερ Γιάρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ζητάει το λόγο, έτσι, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, το ΕΛΚ προτείνει την κυρία Μπεσέρα και την κυρία Ματσόλα. Τις ίδιες δηλαδή αντιπρόεδρους όπως είχαμε και την προηγούμενη φορά. Οι ψηφοφορίε θα γίνουν μία-μία. Λοιπόν, τώρα θέλω υποψηφιότητε, ονόματα δηλαδή, για τη θέση τη πρώτη αντιπροεδρία. Κυρία Στέρα, είπατε μία-μία. Εντάξει. Ωραία. Άλλε υποψηφιότητε, παρακαλώ. Όχι. Κανεί δεν ε, είναι αντίθετο στην εκλογή τη κυρία Εστέρα. Όχι. Καλώς. Ωραία, τότε διαβοής. Ρώσα. Έλα, δεν αισθάνομαι κάπως μόνη εδώ στο βήμα. You was είσαι What was you the second or what? I, need also to call... Πρόεδρος, προσοχή και σε κάτι άλλο. Πρόκειται για το άρθρο 204 του κανονισμού, 204 παράγραφος 1, που λέει ότι πρέπει η ποικιλομορφία του Κοινοβουλίου να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση του Προεδρείου. Πράγμα που σημαίνει ότι το Προεδρείο δεν είναι δυνατό να αποτελείται ούτε μόνο από άντρε, ούτε μόνο από γυναίκε όμω έτσι. Και άρα όλοι οι αντιπρόεδροι δεν μπορεί να είναι του ίδιου φίλου, ούτε και να έρχονται από την ίδια χώρα. Έτσι ήθελα απλώ να σα το πω για να καταλάβετε ότι θέλουμε να ακολουθούμε τον κανονισμό και να λάβουμε υπόψη μας το άρθρο 204. Έχετε λοιπόν πρόεδρο, μια γυναίκα, έχετε μια γυναίκα αντιπρόεδρο, λάβετε το υπόψη σας αυτό. Τώρα που σας ζητάω υποψηφιότητες για την θέση του δεύτερου αντιπροέδρου της Επιτροπής μας, παρακαλώ. Παρακαλώ, ακούω. Πίτερ Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Ματσόλα προτείνω για τη θέση αυτή. Άλλες υποψηφιότητες, παρακαλώ. Ωραία, μπορούμε διαβοής τότε να εγκρίνουμε την δεύτερη αντιπρόεδρο. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, Ρομπέρτα. Ελάτε εδώ κι εσείς στο βήμα. Και τώρα φτάνουμε στη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. Παρακαλώ, Σολεδάδα οι σοσιαλιστές προτείνουν την Μαρλέν Μίτσι. Άλλες υποψηφιότητες παρακαλώ. Διαβοής Δεν Μπορούμε να εγκρίνουμε την ε, τρίτη αυτή αντιπροεδρία, την Μαρλέν Μίτσι. Συγχαρητήρια. Ναι, ελάτε, ελάτε εδώ στο βήμα. Άλλη μια γυναίκα, ναι. Τώρα φτάνουμε στην τελευταία, την ναι. τέταρτη αντιπροεδρία. Παρακαλώ υποψηφιώτες και λάβετε υπόψη σας αυτό που σας είπα πριν, έτσι. Πίτερ, να ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πολύ ευτυχείς να προτείνουμε τον κύριο Τσάκη στη θέση του τέταρτου αντιπρόεδρου. Οπότε έτσι έχουμε και έναν άντρα στο Προεδρείο. Είναι ο υποψήφιος που προτείνουμε. Πρόεδρος, άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν για αυτή τη θέση? Άλλες υποψηφιότητες για τη θέση του τέταρτου αντιπρόεδρου? Ωραία. Ο Πολτσάκη, διαβοής. Εγκρίνεται υποψηφιότητα? Κάλο. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια πάλι. Η θέση σας στο βήμα εδώ καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμη είναι. <laughs> Ελάτε παρακαλώ να καθίσετε εδώ μαζί μας. Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι θα ήθελαν να, να εγκαταλείψουν. Αν είναι έτσι, παρακαλώ βγείτε από την αίθουσα ησύχως για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τη συνεδρίασή μας. I... Συνάδελφοι, τώρα που ψηφίσαμε, έχουμε προεδρείο, πρόεδρο, αντιπροέδρους, οπότε μπορούμε να επανέλθουμε στις εργασίες μας. Ημερήσια διάταξη. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Νοεμβρίου, τις δύο που είχαμε. Τα πρακτικά έχουν κυκλοφορήσει και θεωρούνται εγκεκριμένα. Έχω κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα ότι έχουμε κάποιους καινούριου στο προσωπικό μας και θα ήθελα να στραφώ στην Καραλίνα Αγκαγεύσκα πρώτα απ' όλα και την Μαρέια Σκούντρικ που είναι διοικητική πάλι. Παρακαλώ για να σας δούμε ποιες είσαστε. Ωραία. Λοιπόν, να είσαστε Καλή όλοι με τα κορίτσια, με τις κυρίες. Αν έχετε εσείς πρόβλημα, να έρθετε σε μένα. Θα σας βοηθήσω. Να ξέρετε πάντως ότι δύο αυτές νέες συνάδελφοι γνωρίζουν πολύ καλά τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και μιλούν πολλές γλώσσες. Θα είναι στη διάθεσή σας και θα σας βοηθήσουν πολύ. Καλώς ορίσατε σε μας. Δεν υπάρχει τίποτα για τα διάφορα. Και περνάμε στο σημείο 6 που είναι η αναφορά 0618 όσον αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος στην πόλη Ατσέρα στην περιφέρεια της Καμπανίας, στην Ιταλία. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ, γι' αυτό και θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμέσω, ο κύριος Φερστράτερ. Είναι εδώ? Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως υπήρχε κάποιος προβληματισμός όσον αφορά την μόλυνση των υπογείων αλλά και των υδάτων επιφανείας σε σχέση με κάποιες βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή της Ατσέρα. Και θεωρήθηκε ότι αυτά τα μολυσμένα ύδατα χρησιμοποιούνται για το πότισμα ε, τροφών και ζωοτροφών. Ε, Επίση και το πόσιμο νερό θεωρήσαμε ότι μπορεί να κινδυνεύσει από αυτή την μόλυνση των ε, υδάτων. Και άρα ότι υπήρχε κίνδυνος για τη δημοσία υγεία. Οπότε κατεστεί αποδεκτή αυτή η αναφορά και κατεστεί επίση σαφέ ότι σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο όντως ε, ε, προβλέπεται ότι οι ζωοτροφές αλλά και τα τρόφιμα τα οποία τίθενται σε εμπορία θα πρέπει να ε, υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία ο σχετικός κανονισμός είναι 2002 για τα τρόφιμα και είπαμε ότι εδώ πέρα θα πρέπει δύο ε, ε, PCB και άλλες ουσίες ε, θεωρούνται ότι είναι επικίνδυνες όπως επίσης προβλέπει σχετικά και ο κανονισμός 3.15.93 για τα τρόφιμα και προβλέπει διάφορα τοξικά στοιχεία αλλά αυτό που τα προβλέπει και ο κανονισμός 18.2006 και υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες ουραϊκές τιμές για τα βαρέα μέταλλα που περιέχονται και στην οδηγία 2032. Οπότε, έχουμε και τον κασμό 854 που ορίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα δυνατά μέσα από τις επιχειρήσεις τροφίμων, από τους αγρότες, από όλους, τόσο ώστε να εξασφαλιστεί ότι τρόφιμα και ζωοτροφές δεν θα μολύνονται από διάφορες χημικές ε, ουσίες ε, ή από ουσίε από τη φύση οπότε θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την σχετική υγιεινή άρα δηλαδή όλα τα ύδατα για ποσμό των καλλιεργειών δεν θα πρέπει να έχουν μάλλον αυτά τα ύδατα τα οποία έχουν κάποιο κίνδυνο μόνοι δεν θα πρέπει να σχετίζονται με τρόφιμα και ζωοτροφέ για να μην υπάρχει για δημοσία υγεία είναι σαφέ ότι τα ύδατα που χρησιμοποιούνται για την μεταποίηση, επεξεργασία των τροφίμων θα πρέπει να είναι ποιότητος ε, όπω ε, όπως προβλέπεται από την κοινωνική νομοθεσία. Ζητήσαμε στι τελικέ Αρχές να μας παράσχουν περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το τι ισχύει εκεί στην ε, περιοχή αυτή, τι γίνεται με τη μόλυνση του εδάφους, τι γίνεται με τα υπόγεια φαινικά ύδατα, οπότε να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει μόλυνση ζωοτροφών και τροφίμων και μας είπαν οι αρχές της Ιταλίας ότι υπάρχει κάποιο διάταγμα του 2015. Σύμφωνα με αυτό προβλέπεται ποιες περιοχές σε αυτή την περιφέρεια χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφίμων και για ζωοτροφές. Όταν υπάρχει μεγάλη μόλυνση δεν θα πρέπει αυτό το νερό να χρησιμοποιείται και επίσης οι περιοχές εκεί όπου φυτεύονται ζωοτροφές ή προϊόντα για τρόφιμα θα πρέπει και αυτές να καλύπτονται από αυτές τις διατάξεις. Και έχουμε 82 δείγματα από το 2016 από τρόφιμα και ζωοτροφές, ε, μέλι, αυγά, ζωοτροφές, γάλα και άλλα προϊόντα, τα οποία αναλύθηκαν για, για διάφορες μολυσματικές ουσίες, για κάδμιο, ε, μόλιβδο, πολυχλωρικά ε, διφενόλες και υπολείμματα λιπασμάτων και τελικά θεωρήθηκε ότι υπάρχει συμμόρφωση προς τα όρια του κοινοτικού δικαίου. Δεν ήταν τέτοια ποσότητα αυτές οι ουσίες και όπου βρέθηκαν που να δημιουργούν κίνδυνο. Επίσης, βάσει αυτών των πληροφοριών είπαμε δεν υπάρχει μια σχέση μεταξύ των συμπερασμάτων αυτών των δειγματοληψιών και από την άλλη μεριά μια σχέση με την μόλυνση του περιβάλλοντος. Οπότε με τη βάση αυτών των πληροφοριών που μας έστειλαν, ήταν πολύ εντελέχη, εμείς καταλήξαμε στο ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε δεόντω σε ευθελικέ αργές και ο κόσμος που μένει σε αυτή την περιοχή δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο όσον αφορά την υγεία του. Και σας ευχαριστώ. Ε, εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Please, the floor is yours. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε και συνάδελφοι. Προέρχομαι από την Καμπανία. Και ειλικρινά δεν είναι δυνατόν να θεωρήσω ότι είναι παραδεκτά αυτό μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνη υπέροχα όλα αυτά τα γραφειοκρατικά τα οποία διαβάζω για όλες αυτές τις μολυσματικές ε, ουσίες όλα αυτά που μας έστειλαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι όμως μιλούμε τώρα για κάποια περιοχή μολυσμένη για ένα από τα πιο χτυπητά παραδείγματα μόλυνσης γιατί όμως διότι εδώ υπήρξε παράνομη χρήση τοξικών ουσιών. Ακόμα και πυρηνικά απόβλητα πέσανε εκεί. Και κανένα θεσμικό κανένας υπουργός δεν μπορεί να βρει ένα διέξοδο σε αυτό. Και θα περίμενα από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη να είχε πιο σκληρή αντιμετώπιση, να είναι πιο αποφασιστική. Εδώ πρόκειται περί εκατόμβες, γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα έγγραφα τα οποία προέρχονται από την Ιταλία είναι έγγραφα του 2015. Αυτό σας τονίζω. Τότε δε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο κύριος Ναπολιτάνο ο οποίος κατηγορήθηκε κατηγορήθηκε για συνεργασία με την μαφία, οι οποίοι στην Ατσέρα είχαν αναπτύξει ή της μαφίας τέτοιες δραστηριότητες παράνομης διακίνησης και εμπορίας αποβλήτων. Να, επομένω, πώς προήλθε ο κίνδυνος ζωής. Αλλά παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη τα γεγονότα όχι τόσο σε επίπεδο μόλυνσης, αλλά και σε σχέση με αυτό, αυτή την παράνομη εμπορία, την διεθνή παράνομη εμπορία αποβλήτων. Ερχόντουσαν από παντού, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά περνάγανε από κάποιες επεξεργασίες και κινούντος στην ε, καμπανία και είχαν μπλέξει με τη μαφία όλοι οι σχετικοί εμπλεκόμενοι φορείς. Υπήρχε επομένως τέτοιου είδου συνωμοσία, διαπλοκή μεταξύ ε, της διοίκησης, της κρατικής και της μαφίας. Μα είναι δυνατόν να έχουμε... Κοιτάξτε αυτές τις φωτογραφίες, κοιτάξτε. Πρόκειται ε, για κάποιες φωτογραφίες ζώων, τα οποία εξετράφησαν εκεί. Και βλέπετε ότι γεννήθηκαν με τρία μάτια. Άρα δεν αρκούν αυτοί οι κατάλογοι με τις μορισματικές ουσίες. Αυτά που σας δείχνω είναι πραγματικά περιστατικά. Ζω με τρία μάτια. Σας ευχαριστώ, αλλά παρακαλώ, εάν θέλουμε να έρθει πιο κοντά στον κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε ανάλυση της γραφειοκρατίας των υπαλλήλων της δίκησης. Τη σήμερα ημέρα θα πρέπει να έρθει πιο κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Thank you. Κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Αντινόλφη. Ότι η κατάσταση έτσι έχει. Είναι δραματική. Απλώς να σας πω ότι η αναφορά δεν θα πρέπει να μπει στο αρχείο, να μείνει ανοιχτή. Δεν θα πρέπει να αρκεστούμε στην ε, γελία απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν λαμβάνει υπόψη της με υπεύθυνο τρόπο τις ενδείξεις των όσων έγιναν εκεί στην περιοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σχετικά όλα αυτά. Πέρσι δε είχαμε υποβάλει ερώτηση προς την Επιτροπή όλοι από το κοινό πέντε αστέρων σε σχέση με τις κοινοτικέ χρηματοδοτήσεις που είχαν ε, εκταμιευθεί για τα φυτοπροστατευτικά, τα φυτοφάρμακα τέλο πάντων στην καμπάνια. Ήταν 140 εκατομμύρια, αλλά τελικά απεροφήθησαν και χρησιμοποιήθηκαν, αξιοποιήθηκαν μόνο 8. Άρα χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια για την χρήση αυτών των πόρων. Ε, χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα και να ληφθεί, να λυθεί το πρόβλημα, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αλλά υπάρχει όλη αυτή η νομοθεσία για την υγεία, αλλά θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική, πιο αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι απαράδεκτη μια τέτοια απάντηση προς τους αναφέροντες που έρχονται εδώ σε εμά και θεωρώντας ότι είναι η τελευταία τους καταφυγή, η τελευταία τους ελπίδα για μια λύση. Ευχαριστώ. Δεν έχω κανέναν άλλο στον κατάλογο. Ρικάμπρας. Ευχαριστώ. Και συμφωνώ με τους συναδέρφους. Η αναφορά αυτή είναι από το 2013, πριν από τρία χρόνια δηλαδή. Έχει πέρασει καιρό. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει οι έλεγχοι, οι δοκιμές αυτές που έγιναν, πότε έγιναν. Πρόκειται για δοκιμές που γίνονται σε μόνιμη βάση ή δοκιμές οι οποίες έγιναν και έτυχε όταν έγιναν να πετύχουν καλά αποτελέσματα γιατί ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσετε και σοβαρά σε μόνιμη βάση. Αν δεν γίνονται οι δοκιμές σε μόνιμη βάση, τότε λυπάμαι δεν είναι ικανοποιητική αυτή η απάντηση. Και συμφωνώ με τους συναδέρφους. Θα έπρεπε να μπορούμε να δώσουμε μια σοβαρή και πλήρη απάντηση. Πίτερ Γιάρ. Για να απαντήσω, μάλλον σχολιάζοντα την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ικανοποιεί τη συναδέλφους μου, διότι συζητείται εδώ βέβαια το συνολικό πρόβλημα των απορριμμάτων, ενώ η αναφορά αναφέρεται μονάχα σε ένα τμήμα του προβλήματος αυτού. Γνωρίζουμε ότι η συνολική διαχείριση των απορριμμάτων στην Καμπανία είναι ε, μη ικανοποιητική και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει χρήματα τα οποία δεν απορροφώνται διότι εξακολουθεί να λείπει μια, ένα συνολικό σχεδιασμός για την ε, διάθεση των απορριμμάτων. Η παράκλησή μου είναι, εγώ είχα θεωρήσει ότι μπορούμε να κλείσουμε τη μία αναφορά. Να μην τα ρίξουμε όλα μαζί στο ίδιο καλάθι, το μεγάλο πρόβλημα και το μικρό πρόβλημα. Η αναφορά που συζητούμε εδώ αναφέρεται σε ένα μέρος του προβλήματος της διάθεσης των απορριμμάτων στην Καμπανία. Ας το εξετάσουμε λοιπόν αυτό, εάν η πλουσιφία ζητεί να παραμείνει ανοιχτή, έχει καλώς. Αλλά θα ήθελα να διασωθεί κάπως η τιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε μονάχα στο αντικείμενο της αναφοράς και δεν συζήτησε ολόκληρο το συνολικό πρόβλημα. Ευχαριστώ, Μαρλέν. Ευχαριστώ, Σεσίλια. Δεν επιθυμώ να επαναλάβω τα όσα λέχθηκαν ήδη από τις συναδέλφους μου, δηλαδή ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική για τους αναφερόμενους, που είναι πολίτες, του οποίους εκπροσωπούμε. Η Ελεονόρα Αντινόλφη μας έδειξε τρομακτικές φωτογραφίες ζώων που φαίνεται πως είναι το αποτέλεσμα αυτής της ε, τρομακτικής κατάστασης όλων αυτών των αποβλήτων, απορριμμάτων, τοξικών αποβλήτων που ε, απλώς ε, πετάγονται στην φύση στην ατσέρα. Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε βαθύτερα. Είμαι βεβαία ότι η ζημιά έχει γίνει και στα ζώα και στους ανθρώπους, αλλά μέχρι ότου έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, συγκεκριμένες αποδείξεις. Και εφόσον δεν έχουμε συγκεκριμένες αποδείξεις, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ερευνούμε για να δούμε εάν αν αυτά τα ανάπηρα ζώα που γεννώνται πράγματι είναι αποτέλεσμα αυτής της ρήπανσης και μέχρι να μπορέσουμε να συμπεράνουμε ότι δεν προκαλείται ζημία σε ανθρώπους και ζώα, θα πρέπει να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται ο κατάλογος, δηλαδή εξαντλεί το κατάλογος των ε, αγορητών. Μπορούμε να κλείσουμε εδώ. Ε, ο κύριος Κοζολίνο. Συζητεί το λόγο, κύριε. Εγώ ότι πέραν τη ουσία απάντησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία συμφωνώ θα πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα τη σχετική διάκριση. Ε, γι' αυτό το λέω σχεδόν πάντα στους ε, Ιταλούς συναδέλφους. Είναι πάγιο πρόβλημα αυτό η συλλογή και η διάθεση των απολύτων, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε τι άλλη πρωτοβουλία θα πρέπει να αναλάβουμε ώστε να ξαναπάμε στην ε, καμπανία και να δούμε πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς την κατάσταση και θα ήθελα να στραφώ τώρα προς την συνάδελφα από την καμπανία από το κίνημα των να μην ανακατεύουμε τον ε, πρόεδρο γιατί τα πραγματικά περιστατικά τα οποία επικαλέστηκε είναι αναλυθή. Τίποτα, τίποτα ένδειξη δεν υπάρχουν. Τέτοιου είδου μικροπολιτική είναι παντελώ άχρηστη εδώ για το Κοινοβούλιο τότε εκλαμβάνω ως ε, ε, ένδειξη ενότητας ότι και η ΜΕΝ και η ΔΕΧΗ ζητήσατε να μην μείνει ανοιχτή αναφορά και αυτό και θα κάνουμε θα μείνει ανοιχτή αναφορά και θα απευθύνουμε μια επιστολή προς τις αρχές της περιφέρειας της ε, καμπανίας περί της οποίας πρόκειται και θα τους ενημερώσουμε σχετικώς ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται ε, τους προβληματισμούς των ε, αναφερομένων όσον αφορά τις μολυσματικές ουσίες για τα ε, τρόφιμα, τις ζωοτροφές κλπ. Οπότε θα πρέπει να επανέλθουν οι αρχές και θα πρέπει να μας πείσουν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν το πώς εξελίσσεται η κατάσταση για την διατροφική ασφάλεια στην περιοχή και βεβαίω και όσον αφορά και την υγεία των ζώων. Εγγράφως να μας απαντήσουν. Αυτό θα ζητήσουμε. Συμφωνείτε? Ωραία. Έτσι και θα γίνει. Και τώρα προχωρούμε στην επόμενη αναφορά που είναι 465 και αφορά αυτή την γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας στο Μοντάλτο Ουφούγκο της ε, Ιταλίας. Νομίζω ότι είναι εδώ ο αναφερόμενος ο κύριος ε, Λούπο. Ο Λούπο, είστε εδώ. Α, εδώ. Καλώς ορίσατε. Έχετε εσείς το λόγο. Επομένως, για πέντε λεπτά. Νομίζω ότι έχετε να μας δείξετε κάποιες ε, φωτογραφίες. Έχετε το λόγο κύριε. Από τα μέλη της Επιτροπής να σας ευχαριστήσω προσωπικά αλλά και εκ μέρους της ε, κοινότητάς μου. Ε, δείξατε ευαισθησία και σήμερα τώρα μπορώ να σας σημειώσω για το τι γίνεται σε αυτή την μικρή κοινότητα στην επαρχία της Κοσέντζα. Στις 31 Δεκάτου του 2005 είχαμε αυτές τις, αυτή την εγκατάσταση και αυτό προχθεί από κάποιο διάταγμα του 2002. Από εκεί δόθηκε αυτή η άδεια και σύντομα. Ε, ήταν νεκρό γράμμα τόσο έγραφε αυτό το διάταγμα. Όχι, δεν ανταποκρίνεται αυτή η ηλεκτρική γραμμή στα όσα επιβάλλει ο νόμος για την δημόσια υγεία και η υπεύθυνη τώρα είπαμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις και θα πρέπει να συμμορφωθούν όσον αφορά την απόσταση από τα σπίτια που από πρέπει να περνάει αυτή η ηλεκτρική γραμμή. Υπάρχουν διάφορες προδιαγραφές και είπαμε ότι όπως γίνεται σήμερα είναι πολύ κοντά στα σπίτια αυτά τα σύρματα. Βλέπετε εδώ πόσο κοντά είναι τα σπίτια. Είπαμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα με την ε, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Και οι περιφερειακές αρχές της Καλαβρίας πρέπει να προστατεύσουν την περιοχή αυτή της Λουκέτα όσον αφορά αυτά τα καλωδία υψηλής τάσης. και αυτά τα 400-500 μέτρα δημιουργούν πρόβλημα όσον αφορά την απόσταση. Πρόβλημα στην υγεία των κατοίκων. Και όλα αυτά τα καλώδια και αυτή η μεταλλική πύργη ε, μεταφέρουν πάρα πολύ μεγάλη ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κυρίως για τους ανηλίκους. Έχουμε προσπαθήσει να προσφύγουμε και στις αγγελικές αρχές της περιοχής. Και έχουμε 0,3, 0,4 μικροτέσλα στα 300 μέτρα απόσταση. Αλλά είπαμε ότι αυτά οδηγούν σε βλάβες στην υγεία, σε όγκους που δημιουργούνται στον άνθρωπο. Το αφορά, είπαμε, κυρίως τους ανηλίκους και συμφωνούν οι ειδικοί. Αυτό αφορά και στη δουλειά προς το περιβάλλον. Και είπαμε ότι θα πρέπει να τηρηθούν κάποια όρια όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Ορίστηκε η ιδέουσα απόσταση για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Όμως δεν τηρείται αυτό το οποίο βρέθηκε. με τα σπίτια πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα καλώδια θα πρέπει επομένως να τηρηθεί αυτό το όριο των 0,3 μικροτέσλα. 0,3 έως 0,4. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάτσει να τι ισχύει για αυτή την ακτινοβολία, την ηλεκτρομαγνητική. Περιμένουμε παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προβλήματα, αλλιώ θα γίνουν χειρότερα. Thank you very much and thank you. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. ευχαριστούμε για την αφοσίωσή σας σε αυτό το θέμα. Τώρα στρέφομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον εκπρόσωπή της, τον κύριο Φερστράτερ και πάλι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι έτοιμες σε λίγες ε, μέρες για την Επιτροπή Αναφορών. Όπως πάντως γνωρίζετε ήδη, όσον αφορά την αρμοδιότητα, την κατανομή αρμοδιοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών μελών, όσον αφορά την γενική προστασία του πληθυσμού από ενδυνάμει κινδύνους όσον αφορά την υγεία εξαιτία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, είναι αρμοδιότητα που παραμένει στα χέρια των χωρών μελών. Παρ' όλα αυτά, το 1999 το Συμβούλιο ενέκρινε σύσταση για τον ε, περιορισμό της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η σύσταση αυτή λοιπόν, παρόλο που δεν είναι δεσμευτική, έχει ως πρόθεση να καθοριστεί ένα κοινό πλαίσιο προστασίας από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με οριακές τιμές, προκειμένου να συνεισφέρει στη συνοχή, ενώ οι χώρες μέλη μεταξύ τους έχουν διαφορετικές τιμές ε, ως όριο, οριακές τιμές. Τώρα, οι χώρες μέλη σε τι βαθμό ανταποκρίνονται στις συστάσεις ή όχι. Στη δεύτερη έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2008, η τελευταία έκθεση, διαπιστώσαμε ότι η Ιταλία έχει ένα όριο για την πυκνότητα ροής 10 φορές χαμηλότερο από τόσα όσα συστήνονται στη σύσταση του Συμβουλίου. Μπορείτε βέβαια να ρωτήσετε κατά πόσο η σύσταση αυτή του 1999 ισχύει ακόμα τώρα που είμαστε στο 2016. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια ανεξάρτητη επιτροπή για νεοδιόμενους κινδύνους ή για παλιότερους που επανέρχονται και έχει εντολή για να εκτιμήσει τους κινδύνους από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και πάλι. Βασίζεται η μελέτη αυτή αντικτύπου στα στοιχεία που υπάρχουν όταν εγκρίνεται και η σύσταση. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις νομοδοτήσει αυτές τις χρησιμοποιεί για να δει κατά πόσο τα όσα αναφέρονται στη σύσταση του Συμβουλίου του 1999 εξακολουθούν να ισχύουν ή κατά πόσο πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση. Η πιο πρόσφατη γνωμοδότηση που έχουμε είναι του 2015, σχετικά πρόσφατη δηλαδή, πριν από δύο χρόνια, γιατί είναι από τον Ιανουάριο του 2015, δύο είναι αυτή λοιπόν η γνωμοδότηση, εξέτασε πάνω από 700 επιστημονικές μελέτες και σύμφωνα με τη γνωμοδότηση λοιπόν αυτή το βάρος των ε, επιστημονικών ε, μελετών λέει ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που βρίσκονται κάτω από τα όρια τα οποία συστήνονται στην ε, σύσταση δεν αποτελούν κίνδυνο. Άρα δεν υπάρχει λόγος για να αναθεωρηθεί η σύσταση του Συμβουλίου του 1999 βάσει αυτών. Όπως είπα, στην Ιταλία έχουν εγκρίνει οριακές τιμές 10 φορές πιο χαμηλές από τις αποδεκτές τιμές έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία βάσει της σύστασης του Συμβουλίου. Βάσει λοιπόν αυτών των παρατηρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι δεν υπάρχει βάση για παρέμβαση όπως ζητάει ο αναφέρον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Οι συνάδελφοι τώρα, παρακαλώ. Λάουρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας επισημάνω το εξής. Βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Καλαβρία από πλευράς περιβάλλοντος γιατί ε, σε πολλούς τομείς υπάρχουν οι κίνδυνοι. Ε, θα πρέπει επομένω να αναλάβει επιτέλους δράση η Περιφερειακή Αρχή. Άρα και προκειμένου έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε ένα σωρό μελέτες επιστημονικές, καρκινολογικές, διεθνών ε, φορέων και έχουμε 50 600 Hz ως ε, συχνότητα. Και είπαμε ότι έχουμε αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά ε, πεδία που είναι πάνω από 0,3-0,4 μικροτέσλα, οπότε έχουμε εδώ βλαβερές συνέπειες Τη ακτινοβολίας αυτή που είναι πάρα προσβλεπτική για την υγεία επομένω ε, της περιοχής αυτής από που περνούν αυτά τα καλώδια υψηλή τάσης και θα πρέπει κάτι να γίνει για να εξευρεθεί λύση. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι το να υπάρξει σωστή αξιολόγηση αυτών των επιστημονικών δεδομένων. Θα πρέπει καλύτερα να προστατευτεί το περιβάλλον, η υγεία, και άρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν αυτές οι οριακές τιμές για την ακτινοβαλία σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης για το άρθρο 191 της ε, συνθήκης. Έχουμε επίση και το άρθρο 6 της συνθήκης που αναγνωρίζει κοινοτική αρμοδιότητα ε, επικούρησης των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία της ε, υγείας. Και το θέμα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι τοπικές αρχές για να υπάρξει η, η ουσιαστική εφαρμογή των όσων επιτάσσει η κοινωτική νομοθεσία. Ακριβώς αυτά που γράφει και η αναφορά. Καλούμε επομένω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί, να κάνει ό,τι χρειάζεται, ούτω ώστε να μπορέσουν να πετύχουμε τον στόχο του να σταματήσουν, τέλος πάντων να μειωθούν οι σχετικές επιβλαβείς εκπομπές που είναι τόσο κακές για το περιβάλλον και την ε, υγεία. Ούτε συντρέχει περίπτωση αναρμοδιότητες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο να έχουν ε, αποκλειστική τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να προσέξουν οι Ιταλικές αρχές περισσότερο αυτά τα προβλήματα. Θα πρέπει να πετύχουν κάποια αποτελέσματα χειροπιαστά. Τι γίνεται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για όλη την Ιταλία. Έχουμε άλλωστε και το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος που τα προβλέπει αυτά τα όρια και το άρθρο 191 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Γιάρεκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας συγχαίρω πρώτα για την επανεκλογή σας. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να διευθύνετε τις συζητήσεις με τον ίδιο καλό τρόπο όπως πριν. Οι συνάδελφοι Φως μου μίλησε για μια επιστημονική μελέτη για τα ηλεκτρομαγνητικά αυτά πεδία που θεωρεί ότι έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και άλλων ζωντανών οργανισμών. Πριν από αυτό ακούσαμε όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Επιτροπή έχει εγκρίνει το 99 ορισμένες συστάσεις και πάλι το 2015 και σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αναλυθεί 700 διαφορετικά έγγραφα. Και η ανάλυση αυτή απέδειξε ότι δεν θεμελιώνεται τέτοια ε, επιβλαβής συνέπεια. Υπάρχει λοιπόν μια μελέτη που διαπιστώνει κάποια ε, αρνητικά αποτελέσματα, από την άλλη εκατοντάδες μελέτες που δεν το δέχονται. Εγώ δέχομαι αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι εξέτασε δηλαδή πολύ ε, σε βάθος ε, το ζήτημα αυτό και ε, το ανέλησε ορθά. Είμαι δηλαδή διατεθειμένος να αποδεχτώ τον ισχυρισμό της αυτό. Αυτό είναι το ένα θέμα που έχω να θέσω. Το άλλο το διατυπώνω ως ερώτηση. Τι προέκυψε πρώτα, η αγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ή οι κατοικίες. Θα ήθελα να το μάθω αυτό πριν να διατυπώσω άποψη. Εγώ πάντως Άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουν θεσπιστεί κατόφλια και ότι έχουν αναλύσει πολύ προσεκτικά το θέμα και ότι έχουν την ε, κατάλληλη και επαρκή επιστημονική βάση για να αποδείξουν ότι δεν, ή μάλλον ε, για να καταλήξουν στο ότι δεν αποδεικνύονται αυτές οι ε, δυσμενείς ε, επιπτώσεις. Η κυρία Αλβιόλ. Ευχαριστώ. Θα παρέμβω περισσότερο στο επόμενο σημείο, στην επόμενη αναφορά, αυτό γνωρίζω, αυτή γνωρίζω καλύτερα, αλλά έχει άμεση σχέση με αυτήν, γιατί μιλάμε για μια υψηλή τάση σύνδεση. Έχουν υπάρξει διάφορες αναφορές με το ίδιο αντικείμενο, αυτές οι δύο δεν είναι οι μόνες, κάτι το οποίο μας δείχνει ότι επικρατεί ανησυχία στους Ευρωπαίους πολίτες για αυτού του είδους τις συνδέσεις υψηλής τάσης και για την ακτινοβολία των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Η ανησυχία αυτή υπάρχει λοιπόν μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτομαι. Παρακαλώ, ζητώ συγγνώμη, αλλά μιλάω. Μπορείτε να με ακούσετε. Ευχαριστώ. Μπορώ να συνεχίσω τώρα. Έλεγα λοιπόν ότι προτείνω η Επιτροπή μας, Επιτροπή Αναφορών, να μπορέσει να ζητήσει κάποια μελέτη όσον αφορά την κατάσταση των συνδέσεων υψηλή τάση στην Ευρώπη. Τι τέτοια προγράμματα υπάρχουν, ποιε είναι οι ανησυχίε των πολιτών, τι νομοθεσία διαθέτουμε, τι επιστημονικέ μελέτες διαθέτουμε, γιατί μα έχουν φτάσει πολλέ τέτοιε αναφορές και ίσω θα ήταν φυσιολογικό να υπάρξει κάποια μελέτη από τη δικιά μας την πλευρά για να καταλάβουμε τι ισχύει στην Ευρώπη συνολικά όχι μόνο για μια συγκεκριμένη περίπτωση, να ξέρουμε πόσε τέτοιε συνδέσει ε, πρόκειται να φτιαχτούν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, θα ήταν δυνατό να ζητήσουμε μια τέτοια μελέτη από την πλευρά της Επιτροπής μας. Η Επιτροπή μας θα τη ζητήσει δηλαδή. Πρόεδρος, να απαντήσω αμέσω. Αν θέλουμε μελέτη, αυτό δεν θα το αποφασίσουμε σήμερα, θα έρθει στους συντονιστές και θα συζητηθεί κανονικά στους συντονιστές. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε με αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Ελεονόρα. Ευχαριστώ πολύ. Λαμβάνω το λόγο γιατί θέλω να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Να την διαβάσουμε επίσης προς ενημέρωση και για να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Ένβια. Θα πρέπει δηλαδή κανείς να προβληματιστεί σε αυτή την περίπτωση για το πώς έγινε αυτό το έργο, πώς έγινε η τοποθέτηση αυτών των ηλεκτρικών καλωδίων κοντά στο κέντρο μιας κοινότητας. Όλοι οι επιστήμονες έχουν γνωμοδοτήσει για τη γλυφοσάτη, για τα λοιπάσματα, φυτοφάρμακα και σε εκείνη την περίπτωση είναι διχασμένοι επιστήμονε. Τώρα όμω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άρα θα πρέπει να ισχύσει 100% η αρχή τη προφύλαξης εδώ. Βέβαια πέρασαν 17 χρόνια από το 99, οπότε είχαμε τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη σχετική αξιολόγηση. Πρέπει επομένως να ασχοληθούμε εις βάθος με το θέμα, να μην ανοιχτεί η αγορά να ασχοληθούμε σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και έτσι να ανταποκριθούμε σε αυτά τα οποία θέλουν οι αναφερόμενοι για αυτό που τους ανησυχεί τόσο πολύ με αυτό που γίνεται στην περιοχή τους. Πρόεδρος. Είστε η τελευταία που ζητήσει τον λόγο. Θέλει άλλος... Α, θέλει να μιλήσει ο κύριο Κοτσολίνο. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Συμφωνώ με τα σου είπε η κυρία Εύη. Έχουμε διάφορες απόψεις πολλές φορές από τους επιστήμονες. Όμως εδώ ο αναφερόμενος θέλει κάποια πρωτοβουλία που να μην ε, αφορά το τι γίνεται με όλο το δίκτυο. Θέλει να δούμε τι γίνεται αυτά, τα, τα, τρία χιλιόμετρα, αυτή, αυτό το κομμάτι τέλος πάντων των ε, εγκαταστάσεων, της καλωδίωσης. Άρα, ας προγραμματιστούμε συμπληρωματικά. Τι γίνεται με τον φορέα που ελέγχει το δίκτυο, τι γίνεται με την περιφέρεια ούτως ώστε να υπάρξουν τέτοιες συνθήκες και να λυθεί το πρόβλημα για αυτά τα τρία χιλιόμετρα, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Το είπε η Κομισιόν, το είπε και η τελευταία συνάδελφος για τις επιστημονικές γνώμες που πολλές φορές είναι ε, διαφορετικές. Να δούμε τουλάχιστον όμως εμείς τι γίνεται για αυτό το μικρό τμήμα, το τμήμα του δικτύου που είναι τόσο κοντά στις κατοικίες, πέραν όλων των υπολείπων. Ακριβώς σε εκείνο το τμήμα του δικτύου να υπάρξει παρέμβαση. Ας τα μελετήσει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αναλυφθεί δράση όσον αφορά το διαχειριστή του δικτύου, την τέρνα, και σε σχέση επίσης με την περιφερειακή διοίκηση της Καλαβρίας. you. And uh, Ευχαριστούμε. Δεν uh, τελειώνουμε με πλήρη ομοφωνία, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ένα συμβασμό. Να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, να μην την κλείσουμε. Α, ναι. Πρέπει να δώσω το λόγο στον αναφέροντα. Ναι, είδατε, έχω έναν uh, τμήματάρχη εδώ ναι, αλλά πρώτα ο Γιάρεκ και μετά ο Αναφέρον, πριν ολοκληρώσουμε. Ναι, βιάστηκα πολύ, όπως με την επανεκλογή μου. Βλέπω, παρά την αρχική μου σύσταση, ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θέλουν να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Δεν θα αντιταθώ. Ωραία. Με αυτό το πνεύμα συνεργασίας θα ολοκληρώσουμε σε λίγο, αλλά προηγουμένως το λόγο έχει ο αναφέρον. Έχουμε, είπαμε, αυτό το τμήμα του δικτύου, αυτά τα τρία χιλιόμετρα, τα οποία όπως ε, προέβλεπε το περιφερειακό ε, πρόγραμμα, ε, για το δηλαδή πώς θα τοποθετηθούν αυτά τα καλό στη Λουκέτα. Σχετικά με αυτό σας διευκρινίζω ότι υπάρχουν μελέτες παρά κάποιες αντίθετες υπερχνικές γνώμες. Και είπαν ότι πιο ευαίσθητες κατηγορίες πολιτών, ηλικιωμένοι, παιδιά, ανάπηροι, αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο από την ηλεκτρομαγνητική εκτενοβολία. Okay. I Καταλαβαίνω ότι θέλετε να παραμείνει ανοιχτή. Καλώς, θα παραμείνει ανοιχτή και θα δούμε στη συνέχεια. Βέβαια, μόνο τον Ιανουάριο πήραμε επιπλέον πληροφορίες από τον αναφέροντα. Έφτασα στη γραμματεία δηλαδή και το αντίγραφο αυτών των ε, νέων πληροφοριών της νέας ενημέρωσης στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται πιο πολύ για τεχνικού χαρακτήρα πληροφοριών. Σίγουρα θα τα ξανακοιτάξουμε όλα αυτά και θα τα στείλουμε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Χωρίς να ζητάμε γνωμοδότηση, απλώς ενημερωτικά. Για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Τι λένε και αυτοί. Ωραία. Με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει αν συμφωνούμε, θα επανέλθουμε σύντομα, πιστεύω. Ωραία. Αυτό αποφασίστηκε. Δεν βλέπω αντιρρήσει. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Και σας που ταξιδέψατε από την χώρα σας τόσα χιλιόμετρα και ήρθατε εδώ. Σας εύχομαι καλό ταξίδι πίσω στη χώρα σας. Και τώρα. Επόμενη αναφορά. 1332 το 2016 όσον αφορά το σχέδιο σύνδεσης υψηλής ε, τάσης στην Ισπανία με ηλιοφάνεια. Δεν είναι εδώ η αναφέρουσα που αρχικά θα ερχόταν, ήρθε όμως η Άννα Παλέρμα που την αντικαθιστά και σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ζητούμε από την Επιτροπή αυτή αναφορών να σταματήσει το σχέδιο το οποίο θα περιγράψουμε στη συνέχεια γιατί παραβιάζει πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες έτσι όπως περιγράφονται παρακάτω. Πρόκειται για μια επίθεση που γίνεται κατά του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της υγείας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Πρόκειται για κάτι από το οποίο υποφελείται απλώς και μόνο εργολάβος και κανένας άλλος. Πρόκειται Επίση για την καταστροφή πολλών ειδών που ήδη απειλούνται με εξαφάνιση. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα γραμμή υψηλή τάση πάνω από 400 κιλοβόλτο που ονομάζεται Πλάνα Μορέλια, η οποία έχει να κάνει με χιλιάδε πολίτε που ζουν εκεί σε διάφορα χωριά που είναι μεσαιωνικά, που είναι αναγνωρισμένα παγκομίω όπω η Νικούγια ή η η μορεγια Και εκεί υπάρχουν πολλά αγροκτήματα απομονωμένα σε όλη αυτή την περιοχή. Υπάρχουν ε, οι κάτοικοι που ζουν παραδοσιακά, ασχολούνται με τον αγροτουρισμό, με τα τη αμύγδαλο, τρούφα είναι τα προϊόντα που έχουν εκεί και πολλά άλλα μεσογειακά προϊόντα. Καταστρέφεται και η ύπεθρος, το τοπίο. Καταστρέφεται ένα μεγάλο μέρος της ζωής των κατοίκων του μαεστράδου που θα αναγκαστούν να φύγουν από τα σπίτια τους. Θα γίνει μεγάλη καταστροφή στην υγεία. Το όφελος είναι μόνο ιδιωτικό χωρίς όμως να προσφέρει περισσότερη ενέργεια στην περιοχή. Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο ηλεκτρισμού. Πρόκειται για μια πληγή στην περιοχή, χωρίς κανένα συμφέρον για το κοινό. Το 2016 καταναλώθηκε το μισό πόσο προβλέφθηκε για φέτος. Το δίκτυο αυτό με 86 χιλιόμετρα μήκος θα συνδέσει τους υποσταθμούς Λαπλάνα με την Μορέγια, που ήδη όμως συνδέονται με άλλη γραμμή ψηλής τάσης που βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτήν την οποία θέλουν να φτιάξουν τώρα και είναι παράλληλη με αυτήν. Αρχικά προβλέφθηκε για 132 κιλοβατόρες και στη συνέχεια ενισχύθηκε και έφτασε τις 400. Η πρόεδρος διακόπτη, μιλάτε γρήγορα που σημαίνει ότι οι διερμηνείς δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν επαρκώς και να μεταφράσουν ικανοποιητικά αυτά που λέτε στις υπόλοιπες γλώσσες. Οπότε σας παρακαλώ επιβραδύνετε λίγο για να μπορούν να σας παρακολουθούν. Ευχαριστώ, λέει ο Μιλήτρια. Το δίκτυο λοιπόν αυτό, το οποίο είναι 86 χιλιόμετρα, θα επρόκειτο να συνδέσει τον υποσταθμό Λαπλάνα με εκείνο της Μορέγια, που ήδη συνδέονται με άλλη γραμμή ψηλής τάσεως που βρίσκεται πολύ κοντά από αυτήν που πρόκειται να φτιαχτεί και προχωράει παράλληλα με αυτήν και στην αρχή είχε προβλεφθεί για 132 κιλοβόλτ. Στη συνέχεια όμως ενισχύθηκε και έφτασε τα 400, χωρίς όμως να γίνει καμία μελέτη αντικτύπου. Το νέο ε, σχέδιο δεν προβλέπει την κατάργηση της ε, γραμμής υψηλής τάσης που ήδη υπάρχει, ούτε λαμβάνει υπόψη τη συσσόρευση των επιπτώσεων των δύο αυτών ε, συνδέσεων υψηλής τάσης. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν θα εξακολουθεί να βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην προηγούμενη γραμμή. Η νέα σύνδεση θα έχει 400 τόρες και θα θυμίζει λιγάκι τον ε, πύργο της Βαρκελόνης. Πρόκειται επίσης για υπερβολικό θόρυβο που δημιουργείται στην περιοχή. Η μελέτη λοιπόν αντικτύπου πριν από 8 χρόνια δεν λαμβάνει υπόψη τη διαχείριση της συγχωρήπανσης. Στο πρόγραμμα αυτό επίσης δεν υπήρξε πραγματική συμμετοχή του κοινού και έτσι δεν τηρείται η σύμβαση του άρχους. Η πρώτη πληροφορία για τους ενδιαφερόμενους ήταν η επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης όπου δημοσιεύθηκε εκεί το πρόγραμμα, που απορρίπτει όμως ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει κατακαιρματιστεί επίσης ώστε να εγκριθεί πιο εύκολα και αποφεύγεται έτσι η περιβαλλοντική αξιολόγηση. Οι σοβαρές επιπτώσεις όμως των στέσεων αυτών υψηλή τάση είναι πολύ ε, σοβαρέ, γιατί δυσκολεύουν ε, τον ύπνο, έχουν προβλήματα να προκαλούν στο μεταβολισμό, καρκίνο, λευχαιμία στα παιδιά, ακόμα και αλσχάιμερ. Οι μελέτες που έχουν γίνει ταξινομούν στην κατηγορία καρκινογόνα φαινόμενα της συνδέσεις αυτές, ότι προκαλούν καρκίνο. Όμως η αρχή της πρόληψης αγνοείται σε αυτή την περίπτωση. Παραβιάζεται το άρθρο 191 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επίσης παραβιάζονται και συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης που συστήνουν ε, μετά από πρόσφατες ε, μελέτες οι συνδέσεις ε, αυτές να βρίσκονται 600 μέτρα μακριά από οποιαδήποτε κατοικία. Δεν λαμβάνονται υπόψη λοιπόν οι πλευρές επιπτώσεις. Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά σε κατοικίες. Ο πληθυσμός εκτίθεται λοιπόν σε επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων πολύ πιο ψηλές από αυτές που συστήνονται σήμερα. Επίσης παραβιάζονται οι κοινοτικές οδηγίες προστασίας των ε, φυσικών ε, περιοχών και πλήττονται και περιοχές του Natura 2000, το Λίξ και το Σέβας και περιοχές με ε, διάφορα άγρια πτηνά όπως είναι ο 200 ε, ετός ή αγριόχινα και άλλα ε, πουλιά αποδημητικά και δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις του έργου αυτού στις περιοχές Natura 2000. Επιπλέον, η εκτέλεση του έργου αυτού θα οδηγούσε να κοπούν πολλά δέντρα και φυτά με εκατοντάδες εκτάρια προστατευμένων εδαφών θα καταστραφούν έτσι δάση όπως έγινε και στο παρελθόν. Πρόσφατα, οι διάφορες περιοχές ενδιαφερόμενες της Βαλένθια έθεσαν σε αμφισβήτηση την εκτέλεση του έργου αυτού εξαιτία των αρνητικών επιπτώσεων επί της υγείας, του περιβάλλοντος, του τοπίου και των τουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν ζητάμε να σταματήσει το σχέδιο και εσείς να αποφασίσετε ότι όντως παραβιάζονται οι κοινοτικές οδηγίες που σας ανέφερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ και εσείς κυρία, Αλβιόλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω τις αναφέρουσες. Θέλω να ευχαριστήσω και την πλατφόρμα του Καστεγιών που είναι κατά του έργου αυτού συνδεση υψηλή τάση εξαιτία των καταστροφών που προκαλεί. Έχουμε να κάνουμε με ένα έργο όπου πρόκειται για κερδοσκοπία στην ενέργεια από μια ιδιωτική επιχείρηση που θεωρεί πιο σημαντικά τα συμφέροντά της από την υγεία των πολιτών. Νομίζω ότι τα όσα είπε αναφέρουσα είναι ξεκάθαρα. Αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία, αυτό το έργο υψηλής τάσης που παραβιάζει οδηγίες προστασίας των φυσικών περιοχών, των αγροπτηνών, και των ε, οικοτόπων, την Πανίδα και τη Χλωρίδα. Μιλάμε για ένα έργο που πλήττει επίσης ε, περιοχές της Natura 2000, ε, περιοχές της Υπέθρου, τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε πολύ μικρή απόσταση, μικρότερη από αυτήν που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στόχος δεν είναι να υπάρξει περισσότερη ενέργεια για τις περιοχές αυτές. Όχι, δηλαδή δεν πρέπει να υποφεληθεί η περιοχή από την ενέργεια που θα της προσφέρει το έργο αυτό. Η ενέργεια θα μεταφέρεται μέσα από τις περιοχές αυτές για να πηγαίνει αλλού. Υπάρχουν επιπτώσεις λοιπόν πολύ σοβαρές όπως είπαμε στην υγεία και στο περιβάλλον και καταλαβαίνουμε επίσης ότι αντιβαίνει και στην σύμβαση του άρχους ότι δεν συμμετείχε το κοινό όπως θα έπρεπε, δεν υπήρξε επαρκής διαφάνεια, δεν δόθηκαν επαρκείς πληροφορίες στον κόσμο που κατοικεί στις περιοχές αυτές και ούτε μπόρεσε να συμμετάσχει ο κόσμος γιατί η διαδικασία έγινε αρκετά στα μυστικά. Παραβιάζεται επίσης και η Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 35 που αναφέρεται στην υγεία, και το άρθρο 37 που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι παρκή στοιχεία προκειμένου η δικιά μας Επιτροπή Αναφορών να ανταποκριθεί. Αν μη τι άλλο, πιστεύω ότι η Επιτροπή μας θα έπρεπε να έρθει σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές με μια επιστολή προς την κυβέρνηση της Ισπανίας ζητώντας να σταματήσει το έργο και να ζητήσουμε και περισσότερες πληροφορίες για τις παραβιάσεις στο ΣΕΠΑ, Λίγκο, Νατούρα 2000, τι έγινε με τη συμμετοχή του κόσμου, για το γεγονός ότι ο αντίκτυπος, ε, η μελέτη αντικτύπου έχει γίνει κατακαιρματισμένα, ότι υπήρχε ήδη μια σύνδεση υψηλή τάση και τώρα θέλουν να φτιάξουν μια δεύτερη, οι παραβιάσεις των ε, οδηγιών των ευρωπαϊκών επίσης κλπ. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, ζητάω από την Επιτροπή μας, Επιτροπή αναφορών έρθει σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, πρέπει να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα για να δω τι έχουν να πούνε. Ο Ντάνιελ Φερνάντες Γκόμες έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους αναφέροντες. Ευχαριστώ για αυτά που ακούσαμε και όσα μας είπατε. Τώρα, Όλα αυτά τα στοιχεία έγιναν γνωστά το 2012 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου άρχισε σχετική έρευνα βάσει διαφόρων γραπτών ερωτήσεων των Ευρωβουλευτών. Η έρευνα αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώθηκε κύρια στις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι η ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οδηγία αξιολόγησης αντικτύπου που αναφέρθηκε, που απαιτεί πράγματι τέτοιου είδους έργα από τη στιγμή που πρόκειται για πάνω από 15 χιλιόμετρα διαδρομή πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση αντικτύπου επί του περιβάλλοντος. Επίσης εξετάστηκε και η εφαρμογή της οδηγίας Habitat, νοικοτόπων, που όντως μπορεί να οδηγήσει στο ότι υπάρχουν επιπτώσεις και παραβιάσεις και καταστροφή περιοχών Natura 2000 ή άλλων προστατευμένων περιοχών. Η οδηγία αυτή η Habitat δεν απαγορεύει βέβαια δραστηριότητες μέσα στις περιοχές Natura 2000, απαιτεί όμως οποιοδήποτε σχέδιο, οποιοδήποτε έργο που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ένα άλλο κομμάτι του Natura 2000 πρέπει να περάσει από μελέτη αντικτύπου για τις περιοχές αυτές και βέβαια να προσαρμόζεται στα όσα ισχύουν. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν εφόσον έχουν αυτά τα στοιχεία να επιτρέψουν το έργο, εφόσον δηλαδή έχουν εξασφαλίσει ότι οι επιπτώσεις επί των περιοχών αυτών του Natura 2000 δεν είναι σημαντικά βλαβερές. Επίσης, εφόσον καλύπτονται κάποιες προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα τέτοιο έργο. Δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις, για παράδειγμα, αν ε, υπάρχουν άλλοι λόγοι ε, υπέρ του κοινού. Και τέλος, εφόσον εγκρίνονται αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία συνάδουν με τόσε γίνουν στο Natura 2000. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ξεκίνησε έρευνα, ζήτησε πληροφορίες από τις Ισπανικές αρχές, οι οποίες μας ενημέρωσαν τότε ότι υπήρξε μελέτη αντικτύπου που είχε ξεκινήσει τότε, αλλά που δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα. Η μελέτη αυτή θα λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις του έργου επί των περιοχών Natura 2000. Βάσει αυτών των πληροφοριών λοιπόν καταλήξαμε ότι όσο δεν έχουμε τα συμπεράσματα της αξιολόγησης αντικτύπου δεν υπάρχει παραβίαση. Γιατί μέχρι τώρα όλες οι υποχρεώσεις έτσι όπως προβλέπονται στην νομοθεσία τηρούνται από την Ισπανία. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να σταματήσει την έρευνα μέχρι να υπάρξουν νέοι δείκτες, νέες πληροφορίες που να δείχνουν ότι δεν τηρείται η νομοθεσία. Πρόσφατα μας έφτασαν νέες υπόνοιες από τους αναφέροντες, νέοι ισχυρισμοί που αναλύσαμε και ετοιμάζουμε μια νέα ανακοίνωση που σύντομα θα στείλουμε στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη που δεν σας έδωσα το λόγο αμέσως μετά την αναφέρουσα. Αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε. Και τώρα επιστρέφω στον κατάλογο μιλητών μου. Μαρσελέση, ο κύριος Μαρσελέση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ να υποστηρίξω αυτήν την αναφορά από την Καστελιών. Όπως τα είπε και η κυρία Αλμπιόλ και εγώ έτσι βλέπω τα πράγματα. Τα μεγάλα έργα για άλλη μια φορά αφορούν αυτά τα καλώδια ψηλή τάση και παραβιάζουν τι οδηγίε για το Natura 2000 ε, και άλλε. Παραβιάζεται επομένω το πνεύμα τη ε, νομοθεσία. Αφορά τους εργαζόμενους στην ε, Ήπεθρο και όχι μόνο. Άρα βλέπουμε ότι καταλήγει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα δημοκρατικό έλλειμμα. Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν αφήνεται να συμμετάσχει στη διαμόρφωση της νομοθεσία. Για άλλη μια φορά παραβιάζεται η συμφωνία του άρχους. Και έχουμε ή έχουν κάποιοι τέλο πάντων αυτή την τάση για κάποια έργα να μην κάνουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και έτσι κάνουν κάποια σαλαμοποίηση του έργου, τόσο ώστε να περάσει πιο εύκολα χωρίς την ε, μελέτη των επιπτώσεων. Άρα, να ζητήσουμε από την Ισπανική κυβέρνηση να κάνει τέτοια αξιολόγηση περιβαλλοντικού ε, αποτελέσματος περιβαλλοντικών επιπτώσεων στρατηγικών διαστάσεων, γιατί πρόκειται τελικά για κάτι το οποίο αφορά το ισπανικό δίκτυο. Είναι θέμα ε, ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτά θα πρέπει να την Ισπανία. Τελευταίο σας τονίζω ότι η διοίκηση της περιοχής της ε, Βαλένθια είναι κατά αυτού του έργου και αυτό έχει σημασία για το θέμα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Στερικάβρας στα αγγλικά, στα ισπανικά. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συναδελφοί μου, Αλβιόλ και Μαθελέση και για όσους δεν γνωρίζουν εδώ στην αίθουσα Το ζήτημα των αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια συλλογή ευρωπαϊκών ιστορικών τρομακτικών ε, επεισοδίων. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν και επιχειρήματα κατά του έργου. Πρώτα πρόκειται για μεταφορά ενέργειας και που διεξάγεται από ιδιωτική επιχείρηση. Αλλά θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί εάν το έργο είναι δημοσίου συμφέροντος ή όχι. Είναι δυνατόν, είναι έχει τη δυνατότητα η επιχείρηση αυτή να κατασκευάσει ε, αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος μήκους 86 χιλιόμετρων με εκατοντάδες πυλώνες χωρίς επιρροή στο δημόσιο συμφέρον. Οι αρχές της Βαλένθια έχουν υποψίες, υποψίες ότι τα πράγματα δεν είναι απόλυτα καθαρά. Το 2012 Οπότε τώρα ξανά ξεκίνησε το έργο. Πέρασαν τέσσερα χρόνια από το 2012. Επομένως ξεκίνησε και πάλι, συνεχίζεται αυτό το έργο να καταληθεί η προηγούμενη γραμμή. Επομένως, επιβάλλεται ταχαίως να φρενάρουμε αυτό το έργο και φυσικά να μην ανοιχτεί η αναφορά μέχρι του πετύχουμε το σκοπό μας για το έργο. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, λέει κυρία Σταράς. Πρώτα πρώτα δεν νομίζω ότι τόσο σημαντικό θέμα θα μπορούσε να ε, συζητείται ε, εγκρυπτό. Θα πρέπει κάπως να ρυθμιστεί. Και αυτό το οποίο εγώ θέλω ότι πρέπει να γίνει είναι η Επιτροπή στη συνεργασία με τις αρμόδιες να μας πούν κατά πόσο αυτό το έργο συνάδει προς την ε, νομοθεσία. Αν έχουν γίνει αυτό που πρέπει για τις μελέτες επιπτώσεων, υπάρχουν σχετικές άδειες. Ε, δεν υπάρχουν, θα έχει άδεια το έργο αφού υπάρχουν δυσκολίες προς τούτο, άρα δεν υπάρχει θέμα διοδότησης. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2006 για να διευκολυνθούν τα έργα υποδομής για την εκένωση και μεταφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργεια σε αυτή την ε, περιοχή, την περιοχή του Καστελιών. να ε, καταργηθεί μια απαρχαιωμένη γραμμή, η γραμμή υπαριθμών 1 που περνούσε από εκεί. Άρα δεν πρόκειται περί άχρηστου έργου. Το θέμα είναι κατά πόσο έχουν γίνει όλα νόμιμα σύμφωνα με τις οδηγίε οδηγίες τη μελέτη επιπτώσεων. Μα λέει η Επιτροπή ότι συνεχίζει ανταλλαγή ενημέρωση με τι πανικές αρχέ και θα προβεί στη σχετική επικοινωνία. Ε, περιμένουμε, περιμένουμε να ακούσουμε αν αυτό το έργο είναι σύνομο ή όχι. Να γίνονται όλα δηλαδή νόμιμα. Είναι πολύ απαιτητικέ οι μελέτε ε, επιπτώσεων και σχετική νομοθεσία. Εάν δεν γίνονται όλα όπω πρέπει, δεν δίνεται η άδεια. σχετικη νομοθεσια αν γινονται ολα οπω πρεπει δεν δινεται η αδεια οποτε γι' αυτό και να μην εκτείνει αναφορά και να δούμε τι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτήν την επικοινωνία, ανακοίνωση μετά από την ε, συνεννόηση με τις αυτόνομες ε, διοικητικές αρχές της περιοχής αλλά και τις αρχές της κοινότητας της διοικητικής της Βαλένθια. Μπέατρης, θα είμαι σύντομο συνάδελφε γιατί τα εξήγησαν πολύ καλά και εις βάθος οι συνάδελφοι όλα αυτά τα στοιχεία της αναφοράς. Να προσθέσω όμως το εξής. Βεβαίω και πρέπει να μείνει ανοιχτή η Επιτροπή, γιατί όπω είπε τώρα η Επιτροπή, πρόκειται να προβεί σε ανακοίνωση σχετικά. Οπότε και εγώ ήθελα να πω στον ε, κύριο τη Επιτροπή, ω εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου, ότι πραγματικά εσεί είστε κύριε οι φύλακε των συνθήκων του αν τηρούνται οι οδηγίε, αλλά και όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ο εγγυητής της νομιμότητας. Και όταν μιλούμε για τέτοιες με, μελέτες επιπτώσεων κοινωνικών, περιβαλλοντικών κλπ. η αρχή της ε, πρόνοιας θα πρέπει να ενεργοποιείται. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοι εδώ, μπορεί να μην ε, είναι όλα νόμιμα, μπορεί να έχει καθυστερήσει η μελέτη επιπτώσεων. Επομένως, σε περίπτωση αμφιβολίας, καλύτερα να ισχύσει αυτή η αρχή της προφύλαξης. Πολύ σημαντικό να προστατεύουμε το περιβάλλον. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι να δούμε για ποιο λόγο για ποιο, για ποιο σκοπό επίσης γίνεται αυτό το έργο. Ε, αφού το αναλαμβάνει να το κάνει κάποιος φορέας θα πρέπει να δρά νόμιμα. Αν λοιπόν υπάρχουν εδώ κάποιες σκιές αμφιβολίες ε, τότε θα μπει φρένο. Άρα και εγώ λέω να μην είναι ανοιχτή αναφορά και να παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι απλώ θέμα εδώ επιμελητίας για τη μεταφορά της ενέργειας. Θα πρέπει να προσέξουμε εάν εδώ εφαρμόζεται, αν τηρείται το κοινοτικό δίκαιο. Και εδώ διακυβεύονται πολλά παραπάνω για τον κόσμο. Βεβαίω και έχουν θεμητό συμφέρον οι επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις δημιουργούν πλούτο για τον κόσμο. Όμως όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν νόμιμα από του ιδιωτικού τομέα είτε του δημόσιου ανάλογα σε, από ποιο τομέα προέρχεται το έργο. Ε, ευχαριστώ λέει πρώτος και το λόγο στην κυρία Καμπεθονής. Ε, πρόεδρε, όλα, όλα τα είπαμε και όλοι συμφωνούμε σχεδόν. Όλοι είμαστε στην, στο ίδιο μήκο οπότε στην προηγούμενη αναφορά συζητήσαμε για ένα πρόβλημα ιταλικό. Τώρα είναι ισπανικό. θα βγουν πολλά προβλήματα. Και όλοι έχουμε κοντά μας ένα τέτοιο παράδειγμα όπου ο κόσμος έχει πρόβλημα με τέτοιου καλώδια υψηλής τάσης. Γιατί ακριβώ αυτό παίζεται εδώ. Άρα, δεν είναι ξεκάθαρο να έχουμε εναλλακτικέ, αλλά θα πρέπει να δούμε πώ ακριβώ θα πλαισιωθούν αυτού του είδου τα καλώδια, αυτοί οι πυλώνε υψηλή τάση. Οι μελέτε δεν λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την υγεία. Λένε ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Λένε επομένω πολύ ότι με τα δεδομένα που έχουμε δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει βλαβή, αλλά υπάρχουν, υπάρχουν και οι άλλοι που λένε το αντίθετο, ότι τα πράγματα δεν είναι σίγουρα και μπορεί να υπάρχει κίνδυνο. Οπότε και εγώ αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξουμε. Επίσης, ε, με αυτούς τους πυλώνες υπάρχει βλάβη και στο περιβάλλον και ο κόσμος ανησυχεί και γι' αυτό. Είναι θέμα της κληρονομιάς της φύσης. Προσήγει επομένω στις ερμηνείες που δίνουμε και προσοχή γιατί είπαμε δεν είναι αυτή η περίπτωση μοναδική, δεν είναι μεμονωμένη. Θα πρέπει επομένω η Επιτροπή να ξεκαθαρίσει το εξή. Τι γίνεται με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αυτό το έργο. Η μελέτη έγινε σύμφωνα με τον νόμο ή όχι. γιατί πολλές φορές δεν συνάδουν προς την νομοθεσία οι μελέτες επιπτώσεων. Πολλές φορές τέτοια έργα προχωρούν γρήγορα και συνήθως ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται, περί τίνος πρόκειται. Άρα και αυτό θα πρέπει να βρείτε κύριε της Επιτροπής. Υπήρξε κάποιο είδου ενημέρωση προς τον κόσμο. Υπήρξε κάποια διαδικασία ούτως ώστε ο κόσμο να ξέρει τι γίνεται. Υπήρξε κάποιο είδου διαβούλευση. Νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά ζητήματα και πάρα πολύ κρίσιμα για να δούμε κατά πόσο τηρείται η νομοθεσία και έτσι θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της ως εγγυητής Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας μην είναι η αναφορά επομένως. Και επίσης, πολύ σημαντικό, ότι ζήτησε η δίκηση της περιοχή τη Βαλένθια προς την κεντρική κυβέρνηση να διερευνηθεί εάν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση, αν υπάρχει κάποιο διάδρομος άλλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το έργο. Αυτά να ερευνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τηρήθηκε ο νόμος. Πώς πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Γιατί πολλές φορές ο νόμος είναι απαρχαιωμένος και επιδέχεται παρερμηνίες όσον αφορά αυτούς τους πυλώνες και τα καλώδια ψηλής τάσης. Θα πρέπει όλα αυτά να ξεκαθαριστούν. Άρα, Εάν να εξετάσουμε τι ισχύει με αυτόν τον νόμο, να δούμε αν πρέπει να το αναθεωρηθεί το σχετικό δίκαιο. Πρέπει να ταφούν τα καλώδια, να είναι υπόγεια, τι, τι γίνεται με τη χρήση των διαδρόμων, γιατί αυτό που έχει προτεραιότητα είναι ο κόσμος και όχι τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ, Soledad. Ε, θα επιστρέψω τώρα το μικρόφωνο στην ε, αναφέρουσα για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να διευκρινίσω λίγο για αυτά που είπε η συνάδελφό σα ότι η νέα αυτή γραμμή υψηλής θα αντικαταστούσε την παλιότερη. Δεν ισχύει ότι προβλέπεται η κατάργηση της ήδη υπάρχουσας γραμμής υψηλής τάσης. Όχι. Πρόκειται για συσσόρευση των επιπτώσεων και των δύο αυτών συνδέσεων υψηλής τάσης. Επίσης, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όντως ε, μιλάει για αυτήν την ε, μελέτη επιπτώσεων και θέλουν να την έχουν για να ξέρουν κατά πόσο υπάρχει δεν υπάρχει παραβίαση. Εγώ θέλω να ζητήσω όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ζητήσει από την Ισπανία να σταματήσει το έργο μέχρι τότε. Γιατί δεν μπορεί να έχει προχωρήσει το έργο ο σχεδιασμός του και τα λοιπά να έχει φτάσει ήδη στο στάδιο της εκτέλεσης και της εγκατάστασης. Η ζημιά ήδη γίνεται, η βλάβη ήδη γίνεται σε αυτά τα στάδια. Οπότε ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει το έργο. Έργο στο οποίο δεν συμμετείχαμε και γιατί δεν λήφθησαν υπόψη οι εναλλακτικέ που ήδη υπάρχουν, που θα μπορούσαν να εξεταστούν. Δεν έχει γίνει λοιπόν σοβαρή μελέτη και είναι και ένα έργο το οποίο δεν αντιστοιχεί σε μια πραγματική ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί για το 2016 η πραγματικότητα είναι ότι καταναλώθηκε το ίμιση μόνο από το προβλεπόμενο. Οπότε δεν αιτιολογείται, δεν δικαιολογείται το έργο αυτό για να έχουμε περισσότερη ενέργεια. Και μια άλλη διευκρίνηση που έχει να κάνει και με την προηγούμενη αναφορά. Ναι, υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία... Ναι, ξέρω, μιλάω γρήγορα, λέει η ομιλήτρια. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, λοιπόν, ε, κάνουν ζημιά στην υγεία. Δεν υπάρχουν μελέτες συγκεκριμένες ε, αιτίας αιτιατού, αλλά επιδημιολογικές μελέτες υπάρχουν που μιλούν για καρκίνους ως επίπτωση της ε, έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ευχαριστούμε πάντως που τάχιστα εξετάσατε την αναφορά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αφού εξετάσαμε το θέμα ως κατεπήγον μετά από διαδικαστικό αίτημα των Πρασίνων, δεν λάβαμε το έγγραφο με πλήρη θεμελίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα παράδειγμα όπου θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικές πότε και πότε να μην χρησιμοποιούμε την διαδικασία επίγοντος. Είναι καλύτερα να διαθέτουμε πλήρη ενημέρωση, πλήρη πληροφόρηση και να, παρά να μην έχουμε. Λαμβάνοντας υπόψη το επιχείρημα αυτό. Νομίζω ωστόσο ότι πρέπει να στραφούμε πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού δεν τη επιτρέψαμε αρχικά να εργαστεί. Δικό μα φταίξιμο ήταν αυτό. Δεν του επιτρέψαμε να εργαστούν και να εξετάσουν το θέμα αυτό βήμα προ βήμα. Θελήσαμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται ταχύτερα, ανταποκρινόμενε στο αίτημα των πρασίνων. Μπορούμε λοιπόν να επιστρέψουμε και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει σχετικά με τα όσα εξηγήθηκαν και σε εμά και σε εσά. Να αναλύσετε το θέμα αυτό όσο γίνεται, να επαναφέρουμε το θέμα αυτό στην ημερησία διάταξη και ως Επιτροπή Αναφορών θα στείλουμε επιστολή στην Ισπανική κυβέρνηση, θα ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες, θα στείλουμε βεβαίως επιστολή επίσης στην Περιφερειακή ε, κυβέρνηση της Βαλένσια για να ζητήσουμε και εκεί ενημέρωση. Και θα χρειαστεί να κρατήσουμε βέβαια την αναφορά ανοιχτή σε αυτό το μεταξύ. Νομίζω όμως όλες και όλοι μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν είναι πάντοτε σοφό να σπέβδουμε και να εφαρμόζουμε την διαδικασία κατεπήγοντος, κάτι που δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει πλήρη πληροφόρηση. Ελπίζω ότι Συμφωνείτε. Η αναφέρουσα, κανονικό δεν λαμβάνει τον λόγο πάλι, αλλά έστω θα σα τον δώσω. Αλλά πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λέτε ότι δεν είχατε αρκετό χρόνο σχετικά με την Επιτροπή, ότι η Επιτροπή έτσι δεν μπόρεσε να εξετάσει επαρκώς ε, το θέμα και γι' αυτό δεν ε, μπορεί να το κάνει, οπότε εντάξει, τότε να περιμένουμε. Αυτό είναι αυτονόητο. Πάντοτε όταν συζητείτε μια αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών, πάντοτε προσκαλούνται οι αναφέροντες. Άρα θα προσκληθείτε και πάλι και ελπίζω ότι δεν θα αργήσει η πρόσκληση αυτή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και σας ευχόμαστε καλή επάνωδο στην πατρίδα σας. Για όλες και όλους τους συναδέλφους σας ευχαριστώ. Εδώ τελειώνει η σημερινή συνεδρίαση και θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 το πρωί. Μην λησμονήσετε να φέρετε τις κάρτες ψηφοφορίας και αύριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και σας εύχομαι καλό βράδυ. Οι συντονιστές όμως θα πρέπει να παραμείνουν. Παρακαλώ μην εγκαταλείψετε την αίθουσα και θα συνεχίσουμε αμέσως.